Ε, Καλή σας ημέρα, συνάδελφοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Το πρώτο θέμα της Μέσης Δράξεως είναι η δήλωση της Κομισιόν αφορικά με την τήρηση των εθνικών μισθολογικών συμβάσεων και των μηχανισμών συνταξιοδότησης. Έχουμε ανάμεσα των Επιτροπογιώνες Χάν, τον οποίο και καλωσορίζω. Καλώ ορίσατε κύριε Χάν στο Κοινοβούλιο και στην σημερινή μας συζήτηση. Έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε την δήλωση της Κομισιόν σχετικά με την ανακοίνωση. Ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να ε, ευκρινίσω ορισμένα θέματα σχετικά με το πρόγραμμα διότι υπάρχουν ανησυχίες ευρωβουλευτών λόγω των οικονομικών ε, προϋποθέσεων που προβλέπεται στο ε, πρόγραμμα της Ιρλανδίας και μία νομική διαφορά σχετικά με το το άρθρο 153 της συνθήκης που αποκλεί διατάξεις σχετικά με τις αμοιβέ σύμφωνα με το άρθρο 153 που αναφέρονται εις ε, την ε, ε, ε, στα αμοιβέσια στο κοινωνικό πρόγραμμα. Δεν είναι όμως ένα τέτοιο πρόγραμμα αυτό που απασχολεί την Ιρλανδία. Είναι μια κοινωνική αρρωγή για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και να εμποδίσει την επέκταση της οικονομικής κρίσεως. Γι' αυτό και βασίζεται στο άρθρο 122β 2 ε, του, της συμφωνίας εάν υπάρχει ε, μη κίνδυνος για σοβαρές, ε, σοβαρές δυσκολίες και υπό αυτά σας προϋποθέσεις πρέπει να διευκρινιστούν οι συνθήκες που θα καθοριστούν σαν μέτρο επί οποίο θα βασιστεί το πρόγραμμα βοηθείας προς την Ιρλανδία και βασίζεται στις συνθήκες εφαρμογή του προγράμματος που ε, βασίζεται στα μέτρα που αναλαμβάνονται από το κράτος και πολλές από τις συνθήκες αυτές όπως η μείωση των κατοτάτων μισθών είχαν ήδη προβλεφθεί στο εθνικό πρόγραμμα της Ιρλανδικής κυβερνήσεως που δημοσιεύθηκε 24 Νοεμβρίου του 2010. Ο στόχος ε, των ε, συνθήκων αυτών είναι να μπορέσει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να αποφύγει ανεργία εις ε, τις πιο ευαίσθητες τάξεις. Πρέπει δε να αξιολογηθεί μαζί με την πολιτική δραστηριοποίησης και τις προσπάθειες εξυγχρονισμού του συστήματος διότι ε, βλέπουμε ότι ε, υπάρχει, υπήρξαν πολλές ε, προσαρμογές οικονομικές στους μισθούς διότι υπήρχε ήδη μία μείωση το 2008 και μετά μία μικρή αύξηση το 2009 και η μείωση στους κατώτατους μισθούς μισθούς απλούστατα αποκατάσταση την κατάσταση που υπήρχε ε, πριν από την κρίση. Το άλλο θέμα που αναφέρεται ή στην ερώτηση αναφέρεται ή στις συλλογικές συμβάσεις για να υπάρχει δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα των συνθήκων εργασίας που προσφέρονται στους εργαζόμενους σε όλους τους τομείς, ιδιωτικό και δημόσιο. Η, ε, η Ιρλανδία έχει ε, εγκαταστήσει έναν διάλογο σχετικά με την πολιτική ε, με τις συλλογικέ συμβάσεις από πολλών ετών και αυτό συνέβαλε ή στην επιτυχία της Ιρλανδικής οικονομίας. Υπάρχει η ευκαιρία για τους κοινωνικούς εστέρους να συμμετάσχουν στη διαργασία αυτή και τη χαιρετίζουμε. Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση της Ιρλανδίας θα αναγνωρίσει τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και θα ε, ε, βαστεί το κοινοτικό δίκαιο. Ούτως ή άλλως αυτά δεν αναφέρονται μόνο στην αγορά εργασίας αλλά αποβλέπουν εις το να ανοίξουν ορισμένους κλειστούς τομείς της οικονομίας ε, για να προστατεύσουν την παραγωγικότητα και τους και ε, τους καταναλωτές και να αποκαταστήσουν την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχουν ε, εκπρόσωποι των κομμάτων. Καταρχήν ο συνάδελφος Γκέι Μίτσο, του ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Χθε ένα ε, νέο νόμος ψηφίστηκε στην Ιρλανδία και ε, η νέα κυβέρνηση η οποία αποτελείται από μια συμμαχία ε, τον πρόθυσε ε, και ένας από τους στόχους είναι η επαναδιαπραγμάτευση των προγράμματος προς το παρόν πολλοί στην Ιρλανδία φοβούνται ότι οι προϋποθέσεις που θέτει το πρόγραμμα στήριξης είναι πάρα πολύ περιοριστικές και φοβούνται ότι θα πληρώσουν το κόστος ε, οι πολίτες ε, από τα σφάλματα των ε, τραπεζών. Η νέα κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει τον ε, απόφαση σχετικά με τους κατώτατους μισθούς αλλά σίγουρα θα είναι όλο το πρόγραμμα αυτό θα είναι ιδιαίτερα επώδυνο πολλές από τις δύσκολες συνθήκες ε, που έχουν οριστεί από το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομοδοτικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σίγουρα θα βοηθήσουν στην ε, διευκόλυνση από την κρίσιμη κατάσταση και παρακαλώ την Κομισιόν να καταβάλει προσπάθειες ε, προκειμένου να βελτιωθούν το συντομότερο δυνατόν τα πράγματα και καλό την Επιτροπή να εξετάσει επιγόντως ε, το ζήτημα το των δυνατόν. Η Κομισιόν ασχολήθηκε επίσης με το θέμα της ε, ανταγωνιστικότητας και της εξηγήσεις των δημοσίων οικονομικών. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι δεν είναι δυνατόν όμως με μιας ως διαμαγείας να διορθωθούν όλα τα πράγματα. Πρέπει να λεφθούν υπόψη και οι ευθύνε όλων όσων συνέβαλαν σε αυτή την κατάσταση. Και αυτό νομίζω ότι θα αποβεί προς όφελος της Ευρώπης και της Ευρωζώνης ιδιαίτερα. Παρακαλώ δώστε τα απαραίτητα εργαλεία στους Ιρλανδούς πολίτες. Θα κάνουμε τη δουλειά που μας που προβλέπετε, αλλά δεν ε, μπορούν οι πολίτες της ε, Ιρλανδίας να πληρώσουν μόνο από το, όλο το κόστος. Ευχαριστώ ε, κύριε Μίτσελ, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για 1,5 λεπτό. Ο κύριος Χιούγκς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αυτό το memorandum ζητά περιορισμό των ελάχιστων μισθών στην ε, Ιρλανδία καθώς ε, και περιορισμό των ε, διαφόρων κοινωνικών συνεισφορών. Δεν ξέρω αν είναι αυτό, αυτή η παρέμβαση δικαιολογείται. Το 1-2 μιλά για συμμετοχή και διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και όχι τέτοιου είδους ε, παρέμβαση. δεν μπορεί η Κομισιόν να επιλέγει την ιεραρχία διαφόρων μέτρων με τέτοιο τρόπο. Επίσης επιμένει για την κοινωνική ευημερία προστασία της δημόσιας υπηρεσίας και τους ε, περιορισμούς και τις περικοπές στο δημόσιο τομέα και στις συντάξεις του δημόσιου τομέα. Πώς μπορούν όλα αυτά να δικαιολογηθούν σε σχέση με την συνθήκη που απαιτεί από την ε, Ένωση να περιορίσει τις ανισότητες, να προωθεί το υψηλό επίπεδο απασχόλησης και να αγωνίζεται κατά του κοινωνικού αποκλείσμου. Η μόνη απάντηση απάντηση είναι, Πρόεδρε, ότι αυτά τα, δύο δεν μπορούν, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμφιλειωθούν και να συνδυαστούν και τώρα ως αποτέλεσμα της ετήσιας έκθεσης περί ανάπτυξης όλα αυτά αποτελούν πλέον το γενικό κανόνα. Ο κόσμος όμως απορρίπτει αυτή την ιδέα που βασίζεται μόνο στη λιτότητα. Δεν βλέπουν ποια είναι η κοινωνική πολιτική με χαμηλού μισθού, χαμηλή προστασία προστασία, αδύναμες προδιαγραφές, κοινωνικές προδιαγραφές, καθώς και ε, ψηλότερες ε, μάλλον μεγαλύτερες ηλικίες συνταξιοδότησης. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε ε, για να διαλύσουμε την Ένωση, προχωρήστε, Επίτροπε. Διαφορετικά σταματήστε τώρα. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων για δύο λεπτά το λόγο έχει η κυρία Χάρκιν. Thank President. Mr. Commissioner. Ε, Πρόεδρε, Επίτροπε, εσείς μας λέτε ότι το memorandum αυτό συνεννόησης βασίζεται στο άρθρο 1.2.2, τμήμα 2. Τι γίνεται όμως όταν ένα άρθρο της συνθήκης είναι σε απόλυτη αντίφαση με άλλα άρθρα της συνθήκης. Όπως ρώτησε και ο Χιούζ, πώς αποφασίζουμε για την ιεραρχία, ποιο επικρατεί. Υπάρχει αντίφαση με το 1.5.3, ε, καθώς και με τη sunset clause, την οποία έχουμε έχουμε πολύ συχνά αναφέρει όταν μιλάμε για το Ιρλανδικό πακέτο. Εκεί εφαρμόζονται οι πολιτικές, λέει, και της Ένωσης και δεν θα λαμβάνοντας όμως υπόψη την ε, υψηλή απασχόληση και, την μη, ε, και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και με το θεμελιώδη χάρτη, τι γίνεται όπου οι εργαζόμενοι υποτίθεται ότι πρέπει να ε, κάνουν συλλογικές διαπραγματεύσεις και μπορούν να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους καθώς και να κατέβουν σε απεργία. Πολλοί Ιρλανδοί εργαζόμενοι βλέπουν να βρίσκονται σε τέτοια θέση αυτή τη στιγμή. Πώς αντιμετωπίζουμε την αντίφαση ανάμεσα στα διάφορα αυτά τις συνθήκες λοιπόν. Και άλλη μια ερώτηση, Επίτροπε. Δηλώνεται ότι αυτό το Memorandum of Understanding είναι τελείως αποκλειστικά ευθύνη της Ιρλανδικής κυβέρνησης και ότι η Κομισιόν απλώς ε, το δέχεται. Αν υποθέσουμε ότι έχετε την εξουσία, όπως λέτε, να τα κάνετε όλα αυτά, γιατί δεν κάνετε καμία προσπάθεια να μειώσετε τα μπόνους των τραπεζών, γιατί δεν γίνεται καμία προσπάθεια να εξασφαλίσετε αυτοί που είναι στο πάνω μέρος της ε, μισθολογικής κλίμακας να πληρώνουν το δικό τους μερίδιο, γιατί όταν ε, ε, θέλετε να μειώσετε τα ελάχιστα ημερομήσια, είναι αντιευρωπαϊκά τα αισθήματα που διαπνέουν τους πολίτες μας, βλέπουν τι συμβαίνει βλέπουν πως η Κομισιόν δουλεύει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και αυτό που βλέπουν τελικά είναι ότι περικόπτονται οι ελάχιστοι μισθοί και όσοι ε, πληρώνονται με βάση συλλογικές ε, συμβάσεις ε, πλήττονται από αυτά τα προγράμματα λιτότητας. Μα ποιος αποφασίζει τελικά όμως όταν τα άρθρα της συνθήκης έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πώς ενεργεί η Κομισιόν για να αντιμετωπίσει αυτή την αντιπαράθεση. Εξ των Πρασίνων για 2,5 λεπτά κυρία Κορνέλισεν. Καταλαβαίνω το κατεπήγον από πλευρά Κομισιόν σχετικά με την αντιμετώπιση της ε, οικονομικής κρίσης που απειλεί την σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατανοώ ότι βάλλονται, ε, βάλλονται κανόνες ε, στα, σε κάποια κράτη-μέλη για να αντιμετωπίζουν την κρίση. Αλλά θέλω ότι η Κομισιόν ήταν ιδιαίτερα επιλακτική σε ό,τι αφορά την επιλογή των μέτρων. Αφενός, οποιοδήποτε μέτρο φαίνεται νόμιμο όταν μιλάμε για περικοπή των δαπανών. Όταν η Ιρλανδία ε, μπήκε στον μηχανισμό, αυτό που επηρεάστηκε αμέσως ήταν η μισθή αλλά θεωρώ ότι αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να περιορίζει τους μισθούς. Ε, επίσης ε, δεν κάνετε τίποτα προκειμένου να αυξήσετε κάποιους φόρους στην Ιρλανδία, ιδιαίτερα αυτούς των επιχειρήσεων που είναι ιδιαίτερα χαμηλοί. Και στο κάτω-κάτω μην ξεχνάμε ότι οι περικοπές των δαπανών δεν είναι το μοναδικό ζήτημα το οποίο μπορεί να επηρεάσει τον το χρέος. Γιατί η Κομισιόν βιάστηκε τόσο πολύ να ε, μειώσει τους μισθούς ενώ θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα μέτρα για τις τράπεζες στις οποίες οφείλεται η, κυρίως η κατάσταση. Νομίζω ότι η Κομισιόν δεν αντέδρασε σωστά. Αυτές οι πράξεις και πολιτικές δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να βοηθούν, να βοηθούν το αντιευρωπαϊκό πνεύμα στις ε, χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών εάν η Κομισιόν δείξει την ίδια αποφασιστικότητα όταν πρόκειται για τις κοινωνικές εγγυήσεις που θα πρέπει να παρέχει στους όσους έχουν πληγεί. Ναι, φυσικά ε, επιθυμούμε οικονομική διακυβέρνηση, αλλά θέλουμε για μια ισορροπημένη διακυβέρνηση με την ε, φορολογική βιωσιμότητα. Διαφορετικά οι πιο αδύναμοι θα πληρώσουν το κόστος ε, για ένα ζήτημα το οποίο δεν έχουν καμία ανάμεξη. Εξ ονόματος της Αριστεράς για 1,5 λεπτό ο συνάδελφος Τόμας Χάντλεκ το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η προστατευτική ασπίδα πρόκειτο να προστατεύσει τους ε, ε, πολίτες αλλά τους αφήνει χωρίς άμυνα και πλέον τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται και με τις εθνικές μισθολογικές πολιτικές πράγμα το οποίο είναι ανόητο και ε, δακρύζει κανείς όταν ακούει αυτά τα επιχειρήματα θέματα που δεν είναι καθόλου κοινωνική πολιτική. Είναι απαράδεκτα, δεν είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αντιφάσκει με την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν ήταν ένα περιβάλλον για να υπάρχει κοινωνικό ντάμπινγκ και μείωση των μισθών. Εδώ μιλάμε για μισθούς οι οποίοι θα μειωθούν. Οι μισθοί πρέπει να αντικατοπτρίσουν γνωρίζουν τις συνθήκες της αγοράς. Δηλαδή ε, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι λέγουν τέτοια πράγματα πάσχουν από ε, αχρωματοψία, δεν γνωρίζουν τι σημαίνουν συλλογικές συμβάσεις και ε, δεν προασπίζουν την αυτονομία των πολιτών. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη μισθολογική πολιτική και να ε, ε, ε, υπάρξει μεγαλύτερη κοινωνική ασφάλεια. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρχει μια εξαιρετική τιμωρητική πολιτική μειώσεως μισθών. λεπτό. Πρόεδρε, αυτό ξεπερνά την Ιρλανδία. Πριν από ένα μήνα θύμισα στο σώμα ότι οι συντάξει είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και τώρα ξανά τα ίδια. Χρησιμοποιείται την ίδια γλώσσα περί συντονισμού και μηχανισμών συνταξιδοτικών. Τώρα οι συντάξει ε, συνδέονται πάντοτε με, τις, ε, ε, με τα εισοδήματα. Γίνεται δηλαδή απόπειρα για εναρμόνιση των ημερομισθείων γιατί η συνθήκη λέει ότι τα, η μισθή είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών. Είναι απλό να λέει κανεί ότι η ίδια δουλειά θα πρέπει να πληρώνεται με τον ίδιο μισθό, αλλά όλοι όσοι εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίρνουν τον ίδιο μισθό. Ιδιά σκεφτείτε το κλίμα, το να ζεστάνεις ένα σπίτι κοντά στον αρκτικό κύκλο είναι πολύ πιο δαπανηρό από ότι να ζεστάνεις ένα άλλο ε, στην Μεσόγειο και... Φυσικά ορισμένοι έχουν περισσότερα μετρητά από ό,τι άλλοι. Ε, φυσικά και τα, οι μισθοί δεν μπορούν να είναι ίδιοι η στόχη της Κομισιόν να φτιάξει προγράμματα για να βοηθήσει τα κρατημέλη προς μια ευρωπαϊκή πολιτική ελάχιστων μισθών και τη δημιουργία συνταξιωτικών μηχανισμών είναι κατά των συνθηκών. Αλλά δεν με εντυπωσιάζει πια αυτό. Αυτό κάνει όλη την ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μια εναρμονισμένο συνταξιωτικό σύστημα δεν είναι μόνο ένα όνειρο, αλλά είναι και παράνομο. Αφήστε τα όλα όπως τα έχουν προβλέψει οι συνθήκες. Αυτό θα το αποφασίσει το Westminster στην Αγγλία. Ε, σας ευχαριστούμε και ολοκληρώνουμε με την παρέμβαση των... Τον μία γεγραμμένο συνάδελφων και ξεκινάμε με τον κύριο Μάρτιν. Δύο λεπτά η Ιρλανδία είναι μια τραγική περίπτωση διότι πάντοτε θεωρούσαμε ότι η χώρα αυτή ήταν ένα υπόδειγμα για τα νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως παρόλο που και τότε ε, είχαν προωθηθεί λανθασμένες πολιτικές πράγμα το οποίο δημιούργησε μία φούσκα δισεκατομμυρίων όπου ανεξαρτητοποιήθηκε τόσο πολύ ο τομέα των τραπεζών ώστε δεν υπήρχε πλέον ανταγωνισμός. Και εσείς κύριε Επιτροπέ γνωρίζετε πως οι Αυστριακοί ε, είδαν ε, πόσο καλό ήταν να μετικήσουν στην Ιρλανδία για να αποφύγουν την καταβολή φόρων. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα προς αποφυγή και τώρα όλα αυτά κατέρευσαν. Δηλαδή η φούσκα αυτή απεδείχθη για αυτό που πραγματικά ήταν πράγμα που έλεγαν όλοι στο παρελθόν και πάλι έχουμε μία κατάσταση και όχι μόνο από δικιά μου άποψη όπου για να ανταποκριθεί κανείς εφαρμόζει πάλι ε, μία λανθασμένη πολιτική. Ε, εσείς ε, κύριε Επίτροπε λέγετε ότι ούτως ή άλλως η Ιρλανδία έχει δεσμευτεί αλλά γνωρίζομαι ότι στο τέλος δεν έχουν εναλλακτική λύση τέτοιες χώρες όπως η Ιρλανδία και στη συνθήκη της ε, ε, τη συνθήκη Λισαβόνας ε, είναι κρίμα που δεν την απέρριψαν τη δεύτερη φορά και δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα όχημα το οποίο μπροστά είναι μία πόρσε και από πίσω ε, ποδήλατο. Χρειαζόμαστε κάτι πολύ καλύτερο, χρειάζομαστε σαφή μέτρα αξιολογήσεως, μία οικονομική διακυβέρνηση διότι αυτές οι παλινδρομήσεις δεν θα λειτουργήσουν και θα οδηγήσουν σε μια καταστροφή κάτι το οποίο απευχόμεθα όλοι. Θέλουμε μια Ευρώπη που να λειτουργεί ειρηνικά. Και τώρα το λόγο έχουν οι βουλευτές, ο κύριος Φιλίπ Μπουλόν. Έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με την κρίση και την ε, έκρηξη της ε, φούσκας το δημόσιο χρειάστηκε να παρέμβει σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο και να πλήξει το, τα εισοδήματα αλλά και τα ασφαλιστικά στήματα. Αν η Ιρλανδική κυβέρνηση, η οποία δύσκολα μπορεί να επαναχρηματοδοτηθεί από τι αγορέ προσφύγει στο κονδύλια του Ταμείου Σταθερότητα, τότε θα πρέπει να κάνει αλλαγές στον κοινωνικό και φορολογικό τομέα, ενώ αυτό εμπίπτει στο πλαίσιο της επικουρικότητας. ω γιατρό να πω ότι σε περίπτωση πυρετού δεν χρειάζεται να δίνουμε αντιπυρετικό χωρί να βρούμε ποια είναι η αιτία. Θα πρέπει λοιπόν στην περίπτωση αυτή η χώρα να προβεί σε εξυγίανση των δημοσιονομικών τη για να καλύψει το υπερβολικό χρέος. Αυτό θα βελτιώσει το 10% το το ΑΕΠ τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, οι τράπεζες θα επηρεάσουν την κατάσταση και την ίδια την αξιοπιστία η τράπεζα θα αναγκάσει τον ιδιώτες να διαπραγματευτούν. Και έτσι λοιπόν ρόλη την αρχή της επικουρικότητας η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση ενός μνημονίου που έχει συμφωνηθεί με το Διεθνές Νομιστικό Ταμείο. Αυτό το συμφωνία περνάει από μια μείωση των τιμών χωρίς όμως να ξεχάσουμε τα φορολογικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν. Δεν πρόκειται για μια ανοιχτή ε, παρέμβαση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε θέματα επικουρικότητας, αλλά μια προστασία της ε, σταθεροποίησης των χώρας. Φυσικά χρειάζεται να βοηθούν τόσο η Ιρλανδία όσο και άλλα κράτη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, κάτι το οποίο προστατεύει και εμάς, αλλά όχι πάση θυσία. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες υποχρεώσεις του. Ευχαριστώ κύριε Μπουλό. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία και να σας πω ότι αν διαβάζετε τόσο γρήγορα οι διερμηνείς αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και θα ήθελα λοιπόν μια που είμαι αρμόδιος για θέματα πολυγλωσσίας να σας πω ότι στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου εξετάζουμε ένα σύστημα διαφορετικό αυτό που έχουμε τώρα. Το υπάρχει ένα σύστημα όπου ο διερμηνέας μπορεί να ενημερώσει τον πρόεδρο που ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό των βουλευτών, ρυθμό των ομιλιών. Εμείς θα φροντίσουμε να αλλάξει το σύστημα και έτσι να, να βοσβήνει ένα φωτάκι στο έδρανό σας ώστε να μην χρειάζεται να σας διακόπτει ο Πρόεδρος αλλά να γνωρίζετε ότι δημιουργείται πρόβλημα στους διερμηνείς διαβάζοντας με τέτοια ταχύτητα. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα χρειάζεται από εδώ και στο εξή να διακόπτει ο Πρόεδρος και να σας το υπενθυμίζει. Ο κύριος Προήνσιας Ντερόσα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το Μνημόνιο Συνεννόηση όσον αφορά τα θέματα της αγοράς εργασίας βασικά ε, που στηρίζεται σε μια πολύ απλή οικονομική θεωρία ότι κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά θα καθαρίσουν την αγορά όπως λέει, δηλαδή θα εξαφανίσουν την ανεργία. Μα αυτό είναι ανοησία. Δεν υποστηρίζεται από την πράξη στο έδαφο, στη επιτόπου. Ε, πέρυσι έγινε μια έρευνα που λέει ότι οι εταιρείε ε, προτιμούν τις απολύσεις γιατί κοστίζουν λιγότερο. Αυτή είναι η βάση. Γιατί είχαμε τόσες απολύσεις και μείωση των μισθών. Εγώ θα έλεγα απλώ στην Κομισιόν να, να, να κοιτάξει τίποτα άλλο, να κοιτάξει τη δολίτσα τη και να αφήσει ήσυχη την Ιρλανδία για του μισθού. Εμεί έχουμε μακρά παράδοση ε, συλλογικών συμβάσεων και είναι η βάση για το γεγονό ότι δεν υπήρξε βία στου δρόμου στην Ιρλανδία. Γιατί ακριβώ η κοινωνική εταίροι και η κυβέρνηση έκαναν τι δικέ του ρυθμίσει για να ρυθμίσουν την αγορά εργασία και να εξασφαλίσουν ότι μπορούμε να έχουμε κάποια ελπίδα ανάκτηση από τη σημερινή κρίση, ανάκαμψη μάλλον από τη σημερινή κρίση. Κομισιόν και τα πέτρα της δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν την πρόοδο στην Ιρλανδία, αλλά ε, δεν κάνει καν αυτό που είχε υποτίθεται ότι θα κάνει. Ε, να βοηθήσει δηλαδή την ανάπτυξη της οικονομίας στην Ιρλανδία. Δεν ανάπτυξη της οικονομία ε, παρακμάζει και τα θέματα που σχετίζονται με την ε, αγορά εργασίας θα πρέπει να αφαιρεθούν. Η Ιρλανδική κυβέρνηση της οποίας είναι μέλος του δικό μου κόμμα έχει ήδη δηλώσει ότι θα αντιστρέψει την ε, περικοπή ελάχιστου μισθού. Ε, μπορεί να μην σας αρέσει αλλά αυτό θα γίνει. Μπορείτε να είστε και βέβαιος ότι η απόπειρά σας να παρέμβετε με το νόμο περί απασχόλησης που ισχύει εδώ και 50 χρόνια και προσπαθείτε εσείς αυτό να, να επηρεάσετε δεν θα το καταφέρετε γιατί η κυβέρνησή μας ακριβώ παίζει το ρόλο που πρέπει να παίξει να εξασφαλίσει την ειρήνη την ειρήνη ανάμεσα στους εργαζόμενους. Σας παρακαλώ πολύ να ολοκληρώσετε γιατί έχετε ξεπεράσει το χρόνο. ευχαριστώ. Ενάμιση λεπτό η κυρία Φιγερέδο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η τάση που διαπιστώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, να πιέζονται τα κράτη-μέλη, να υποβαθμίζονται οι μισθοί ή να πιέζονται, συμπιέζονται οι εργαζόμενοι ώστε όλα ένα και μεγαλύτερα, περισσότερα πλούτη να αποκτάνε οι εκπρόσωποι του καπιταλισμού. Είναι παράλογα τα κριτήρια του Συμφώνου σταθερότητα με τις προτάσεις τη υποτιθέμενη οικονομική διακυβέρνηση και το Σύμφωνο ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, μείωση ακόμα μεγαλύτερη των μισθών, αποσύνδεσή του από την ε, τιμαριθμική αναπροσαρμογή και γενικά περιορισμό των κοινωνικών και εργατικών δικαιωμάτων αυτό που συμβαίνει ήδη σε κάποιες χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί μειώνονται οι μισθοί, μειώνονται οι συντάξει, ακόμα και οι πιο χαμηλέ, που είναι κάτω και από τη γραμμή τη φτώχεια. Στην Πορτογαλία έγινε μια περικοπή του, ελάχιστου εθνικού μισθού που προεβλεπόταν για φέτο. Θεωρήθηκε ότι ήταν πάρα πολύ υψηλό το ποσό των 500 ευρώ το μήνα και αποφάσισαν να κόψουν 15 ευρώ. Και μην σα πω πόσα παίρνουν οι ε, γυναίκες οι εργαζόμενε. Όσον αφορά τους άντρες, ε, ε, αυτό καλύπτει το 60% των εργαζόμενων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο, μαζί με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, στην ουσία ε, επιτείνει τις ε, ανισότητες, ε, υποβαθμίζει την εργασία, την νομοθεσία, την εργατική και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό και εμείς θέλουμε να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας στους νέους επαγγελματίε που θα αγωνιστούν τις επόμενες εβδομάδες, ήδη από το Σάββατο 12 Μαρτίου, μετά στις 19 Μαρτίου έχει διοργανωθεί μεγάλη μεγάλη ε, διαδήλωση της ε, ΤΕΜΠΕ στη Λισαβόνα και που θα διαμαρτυρηθεί κατά αυτών των αντικοινωνικών ε, μέτρων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάρτς Πίτερ Μάρτιν θέλει να σας θέσει ερώτημα. Δέχεστε? Έχω μία ερώτηση προς εσάς. Μετά από τα όσα μας είπατε θα μπορούσατε να μας αναφέρετε ποια είναι η στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πορτογαλία των πολιτών. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν, έχει αλλάξει η αντιμετώπιση τους, έχουν υπάρξει εξελίξεις. Ποιο είναι το γενικότερο συνέστημα στην Πορτογαλία. Διότι η Πορτογαλία παρουσιάζει κάποιες αναλογίες ε, σε σχέση με την Ιρλανδία είχατε κι εσείς ε, μία φούσκα στον τομέα των ακινήτων όπως συνέβη και στην Ιρλανδία. Έχετε τρία δευτερόλεπτα για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ. Είναι ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Ως προς αυτό είναι προφανές ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές δημιουργούν μεγάλη αποστροφή και επαναστατικό πνεύμα και στην Πορτογαλία. Και γι' αυτό και την επόμενη εβδομάδα ε, θα κατέβουν όλου του δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά αυτής της ε, πολιτικής και στις 19 ε, θα κάνουμε στην Λισαβόνα διαδήλωση της Ομοσπονδίας Εργαζομένων, Γενικής Ομοσπονδίας Εργαζομένων της Πορτογαλίας. Η χώρα μας βρίσκεται σε ύφεση και ο κόσμος ζει όλο ένα και επιχειρότερα. Οι ανισότητες επιδεινώνονται και η φτώχεια επιδεινώνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, ο Πρόεδρος διακόπτη. Να τέλειωσε ο χρόνος σας. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Μαρίτα Ουλσκογ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είπατε ότι για να... η επιβολή μάλλον ε, κάποιων ε, αποφάσεων και κανόνων ε, μπορεί να ρυθμίσει κάποια ζητήματα και να βρεθούν λύσει σε προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα οποία αναφέρατε θεωρώ πως παραβιάζουν τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για ένα μονομένο φαινόμενο που πλήττει μόνο την ε, Ιρλανδία. Πλήττει και άλλες χώρες διότι επηρεάζονται οι μισθοί και όχι μόνο οι συλλογικές συμβάσεις και διαπραγματεύσεις. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξουν νέοι και κανόνες διότι τα κράτη βλέπουν ότι σε επιβάλλεται ένα δικτάτ άνωθεν που επηρεάζει τους πολίτες ε, στην καθημερινότητά τους. Και αυτό το οποίο δημιουργούμε είναι ένα κύμα δυσαρέσκειας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ στο Κοινοβούλιο Ξέρω ότι πολλοί έχουν αρχίσει να ψαρεύουν σε αυτά τα θολά νερά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Μαρίτα. Το λόγο για ένα λεπτό έχει ο κύριος Γιόγκο Κορνέλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. την στις κάτω χώρες υπάρχουν ελάχιστοι οι οποίοι φαντάζονται ότι συζητάμε στις Βρυξέλλες για τους μισθούς τους και τα ημερομίσθια τους. Ε, βεβαίως ε, ξέρω ότι θέλετε να καταργηθούν ε, οι τιμαριθμικές προσαρμογές των μισθών και να συνδυαστούν με μία αύξηση της παραγωγικότητας. Όταν όμως μιλάμε για ένα ελάχιστο ε, ευρωπαϊκό μισθολόγιο υπάρχει σιγή. Θέλουμε να πληρώνονται σωστά και αξιοπρεπώς οι εργαζόμενοι και εγώ απασχολούμαι και ανησυχώ όχι μόνο για τους εργαζομένους αλλά και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που προωθούν τα συμφέροντα των κερδοσκόπων και ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να φροντίσει να ληφθεί υπόψη σαν κάποιος ο οποίος φροντίζει τους εργαζομένους. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό κύριε Ράπτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Χάν, μας είπατε μία συνταγή. Μία συνταγή που λέει δύο πράγματα. Να καταργήσουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας από τη μια μεριά και να κατεβάσουμε και άλλο, να μειώσουμε και άλλο τους κατώτατους μισθούς. Αυτή τη συνταγή την δίνεται συνεχώς σε κάθε ασθενή. ένας από τους ασθενείς είναι η ελλάδα. ήρθατε πρόσφατα εκεί κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης που διοργάνωσε το σοσιαλιστικό κόμμα. είδατε και αισθανθήκατε την κατάσταση που επικρατεί και το ερώτημα που θέτω είναι η συνταγή αισθανθήκατε ότι στην ελλάδα έπιασε τόπο; γιατί εγώ που είμαι από εκεί και που προέρχομαι από το σοσιαλιστικό κόμμα που σήμερα κυβερνά τη χώρα και κάνει ό,τι μπορεί για να τη βγάλει από την πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία την έριξαν οι κυβερνήσεις της δεξιάς έχει αναγκαστεί να βάλει νερό στο κρασί της να βάλει νερό στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αλλά ακόμη δεν βλέπουμε αποτελέσματα λέτε ότι το κάνετε για τον ευρωπαίο πολίτη για τον καταναλωτή μα αν ο καταναλωτής πάρει λιγότερο μισθό δεν θα έχει να ξοδέψει άρα δεν θα βοηθήσει την ανάπτυξη. το ξέρετε καλύτερα από μένα ότι είναι φαύλος κύκλος. γιατί επιμένετε να δίνετε μια συνταγή που δεν οδηγεί πουθενά αλλού παρά μόνο στην κατάργηση της αξιοπρέπειας του εργαζομένου μια συνταγή που οδηγεί στο να μην υπάρχουν αξιοπρεπείς και διατηρήσιμες θέσεις εργασίας. παρακαλώ πολύ εκτός από τους οικονομικούς δείκτες βάλτε και δείκτες señora, κοινωνίας... Κυρία Ράπτη, ξεπεράσατε κατά πολύ το χρόνο ομιλία σας. Η κυρία Γιούτα Στέινμπρουκ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πολλές φορές θεωρώ ότι θα έπρεπε να εφαρμόσετε όλες αυτές τις συνταγές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δείτε τι συμβαίνει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Διότι εγώ έχω την εντύπωση ότι μένετε σε έναν γυάλινο πύργο μόνοι σας και δεν λαμβάνετε υπόψη τους συνταξιούχους, τους ε, μισθωτούς, τους εργαζομένους και αναλαμβάνετε ό,τι αρμοδιότητες σας αρέσει Ήδη πέρυσι τον Οκτώβριο, 19 Οκτωβρίου, έκανα μία ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μου είπαν ότι η μισθή και η κατώτατη μισθή είναι υπόθεση των κρατών μελών. Για διαβάστε το. Δεν είναι δυνατόν τώρα να ε, ε, απαντάτε έτσι από τη μία πλευρά και όταν σας συμφέρει αλλάζετε κατεύθυνση, διότι αυτό όντως ε, δυσαρεστεί πολύ τους Ευρωπαίους και οι συνάδελφοί ε, ε, πολύ σωστά σας τα είπατε. Επεμβαίνετε στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, επεμβαίνετε στους εργαζομένους. Αυτοί που δημιούργησαν την κρίση πρέπει να πληρώσουν και τα σφασμένα. Ευχαριστώ πολύ Γιούτα. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Βλίνκεβιτσουίτε Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπό συνθήκας οικονομικής κρίσεως τα κράτη πρέπει να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και οι δυνατότητές τους είναι όμως διαφορετικές εάν μιλάμε για να ε, επιλύσουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την κρίση. Πρέπει να ισοσκελίσουμε τους προπολογισμού, να λύσουμε τα προβλήματα. Πρέπει όμως αυτό να γίνει εις βάρος αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη μέσα στον πληθυσμό, διότι ότι θα έπρεπε, είναι ανάγκη να μειώνουμε και τους μισθούς. Μιλήσατε για το, τη συμφωνία με την ε, Ιρλανδία αλλά και στην ε, Λετωνία ζητήσατε να μειωθούν οι συντάξεις πράγμα το οποίο έπραξε η χώρα αλλά ε, το συνταγματικό μας δικαστήριο ακύρωσε την πράξη αυτή ως αντίθετη προς το Σύνταγμα και ως εκ τούτου θα έπρεπε να αξιολογήσει και στην Ιρλανδία τις κοινωνικές επιπτώσεις. Ολοκλώνουμε αυτόν τον γύρο μιλών με την παρέμβαση της αδέλφου Ρένιερ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Χάν. Ήδη ε, υπάρχουν πολλά προβλήματα και τώρα στους πολίτες βάζετε ένα βαρύ σακίδιο στην πλάτη και τους, λένε να τρέχετε, να ε, τους λέτε να τρέχουν πιο γρήγορα. Αυτά είναι ε, περί ορισμένες κινήσεις οι οποίες δεν παρουσιάζουν καθόλου μακροοικονομικό συντονισμό. Επίσης ήδη βάζετε διαφορετικά μέτρα και σταθμά για την φορολογία των χρηματιστηριακών πράξεων. Οπότε εγώ αντιλαμβάνουμε τελείως διαφορετικά την οικονομία αγοράς. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες ε, αποκεντρωμένες συλλογικές συντάξεις, ε, ε, συμβάσεις. Πρέπει να υπάρχει σύγκληση των μισθών και όχι από Δηλαδή έπρεπε να γίνει ε, το αντίθετο και γι' αυτό συμφωνώ με αυτά που είπε η συνάδελφο Στάινμπρουκ. Πρέπει να επέμβουμε εκεί που πραγματικά δημιουργήθηκε η κρίση από πλευρά νομοθετική και να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που δημιούργησε η κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα περνάμε στον γύρο του Κάτσου και έχουμε έξι συναδέλφους ε, που έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Μπατσέσκου έχει το λόγο. Ένα λεπτό έχει τη διάθεσή σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά το θέμα του κόστους ε, του εργατικού δυναμικού και της παραγωγικότητας νομίζω ότι θα πρέπει να δίνουμε λιγότερη σημασία σε αυτούς τους δείκτες. Η παραγωγικότητα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εξαρτάται από το ποσό του κεφαλαίου το οποίο διατίθεται και τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ Γερμανίας και Ρουμανίας θα έλεγα διότι έχουν διαφορετικές οικονομικές πολιτικές ε, από πάντα. Αυτές οι διαφορές λοιπόν δεν μπορούν να καλυφθούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η χώρα μου καταβάλει προσπάθειες για αλλαγές στον συνταξιωτικό τομέα και το θέμα της κοινωνικής ασφάλειας. Φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ηλικία συνταξιοδότηση με την δημογραφική εξέλιξη. Μια πραγματική πολιτική στον τομέα των συνταξιοδοτήσεων έχει και αυτή την επιρροή τη στον το οικονομικό τομέα. Ευχαριστώ. Ο κ. Κούρτας έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατανοώ πολύ καλά την αρχή της επικουρικότητας, αλλά θεωρώ πως οι συντάξεις ε, εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Λόγω της ε, οικονομικής ε, κρίσης ε, που αντιμετωπίζουμε της γύρανσης του πληθυσμού και της αύξησης του βιωτικού επίπεδου αλλά και του προσδόκιμου ζωής δημιουργούν διάφορα προβλήματα με τα κοινωνικά ταμεία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Εμείς στην Ευρώπη ξέρουμε έχουμε τους πολίτες οι οποίοι κατά πολύ εξαρτώνται από αυτά τα κοινωνικά συστήματα το ζήτημα των ιδιωτικών της ιδιωτικής ασφάλισης ε, για μας, για τη Ρουμανία, αποτελεί ένα πολύ μακρινό όνειρο για τους ε, πολίτες μας. Ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση θα ήταν να γίνει μια συγκριτική ανάλυση των ε, συνταξιδοτικών συστημάτων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κυρία Μαρίζα Ματίας έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε. Εδώ συζητάμε για προτάσεις για τους μισθούς και για τις συντάξεις και το μήνυμα που μπορούμε να πούμε για αυτές τις προτάσεις είναι ότι ειλικρινά είναι άδικες. Άδικες και πρόκειται για συνταγές που έχουν ήδη δοκιμαστεί και έχουν αποτύχει αυτό που συμβαίνει στην Ιρλανδία, στην, ε, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία και δεν ξέρω και σε πόσες άλλες, ε, άλλες χώρες γιατί είναι μια λυσίδα χωρίς ε, τέλος. Είναι διαφορετική η κατάσταση και σε ορισμένε χώρες όμως υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία. Ποιο είναι αυτό το κοινό στοιχείο είναι η μείωση της αξίας της εργασίας υπέρ του κεφαλαίου. Κάτι ακόμα που, είμαστε, που είναι κοινό είναι ότι αυτό που πληρώνουν την κρίση είναι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι και μια ολόκληρη γενεά επισφαλών εργαζομένων που δεν έχουν καμία εγγύηση. Ε, και θα ήθελα να τελειώσω, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και να οδηγούμε τον κόσμο στη φτώχεια. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε, Μαρίζα. Πάει ο χρόνος. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει κυρία Γιάκον Ευχαριστώ. Προς το παρόν η τάση που υπάρχει στην Ευρώπη είναι ε, λαϊκίστικη δεξιά. Και αυτό σημαίνει ότι η κοινωνική Ευρώπη χάνει προς όφελος ε, της ε, δεξιάς και δεχόμαστε επιθέσεις σε όλα τα επίπεδα, σε μισθολογικές συμβάσεις, σε συλλογικές διαπραγματεύσεις κλπ. Όλα αυτά φυσικά δεν βοηθούν σε τίποτα την επίλυση της κρίσης, οδηγούν σε ύφεση. Για μια ακόμα φορά τίθεται ένα αφιβόλο η κοινωνική Ευρώπη. Θέλουμε να βελτιωθούν τα πράγματα, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας ε, και ασφάλισης ε, των ε, πολιτών μας. Ευχαριστώ κύριο Ρούμπικ, έχει το λόγο. Δυστυχώς η Ιρλανδία δεν είναι η μόνη χώρα η οποία πλήττεται από αυτή την κατάσταση. Υπάρχει και η Ελλάδα και η Λετωνία όπου χρειάστηκε να υποστούμε τις επιπτώσεις όλων των μέτρων που επέσυρε η τραπεζική κρίση. Η κατάσταση στη Λετωνία είναι όπου οι μισθοί έχουν μειωθεί κάτω από το επίπεδο επιβίωσης και οι κατώτατοι μισθοί οι οποίοι είναι αφορολόγητοι και αυτοί έχουν μειωθεί. Οπότε η Λετωνία έχει χάσει το 1 έκτον του πληθυσμού της πολλοί ε, μετακινήθηκαν στο εξωτερικό ε, και σας ζητώ να σώσετε την Λετωνία ε, χωρίς να συνδυαστεί η προσπάθεια αυτή με δρακόντια μέτρα διότι λέγουν ότι υπάρχουν ακόμη αποθέματα για την διάσωση των της χώρας αλλά όχι για τους ε, ανθρώπους. Τελευταίος και ο κ. Ζαντένης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω την ε, ε, στήριξή μου στον κύριο Ρώσα διότι δυστυχώς οι ε, προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αποβλέπουν στο να πληρώσουν οι εργαζόμενοι τα σπασμένα για αυτά, τις καταστάσεις που δεν προκάλεσαν και υπάρχει και μία μείωση μείωση ε, των συντάξεων συνδυάζοντα τις με την ε, προσμονή επιβιώσεως και η ε, τη μαριθμική προσαρμογή ε, των ε, ε, μισθών ή τον πληθωρισμό στη χώρα μου, στο Βέλγιο. Άρα τώρα θα έπρεπε ο Επίτροπος να ακούσει το μήνυμα των εργαζομένων της Ευρώπης για να μην δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των θεσμών και των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νταρθέν. Ολοκλώθηκε ο γύρος των αγοριτών που ζήτησαν το λόγο με βάση το Catch the Eye και θα ολοκληρώσουμε με την παρέμβαση του Επιτρόπου Χάν, ο οποίος ε, θα σχολιάσει τα, ε, τις παρατηρήσεις που έγιναν. Κύριε Χάν, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους ε, όσοι συμμετείχαν στην συζήτηση και θα φροντίσω να λάβω σοβαρά υπόψη μου τις παρατηρήσεις τους. Να πω μερικά λόγια αρχικά σχετικά με τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου. Φυσικά και αναγνωρίζουμε την ε, σημασία αυτού του κοινωνικού διαλόγου και το, στο πλαίσιο των βιομηχανικών ε, σχέσεων ε, και είναι ένας διάλογος τον οποίο προωθούμε σε, όλες τα, σε όλα τα κράτη-μέλη. Ο Επίτροπος Ρεν τελευταία συνάντησε τους ευγεφαλείς ε, των κομμάτων στην ε, Ιρλανδία για να διαπραγματευτούν ε, το πρόγραμμα. Φυσικά θα συνεχίσουμε μέσω μιας αποστολής του μήνα Μάιο αλλά και περαιτέρω. Η Κομισιόν δεν επέβαλε στην Ιρλανδία να μειώσει το κατώτερο, τους κατώτερους μισθούς. Αυτή είναι μια απόφαση της ε, Ιρλανδικής κυβέρνησης ε, στο πρόγραμμα ανάκαμψης για μια ακόμα φορά σε αφορά την ε, νομική βάση αυτή είναι το άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού 407-2010 που προσδιορίζει τον μηχανισμό σταθεροποίησης και το άρθρο 2.2 της απόφασης του 2011 77 Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, δημοσιονομική στήριξη της Ιρλανδίας που αναφέρεται στο άρθρο 122 παράφος 2 της ε, συνθήκης σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι το μνημόνιο κατανόησης ε, συγκεκριμένων οικονομικών πολιτικών που θίγουν πολλές πτυχές και που συνδέεται με την κοινωνική πολιτική δεν ε, θέτει αμφιβόλο την νομική βάση της πράξης. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία αντίφαση ούτε με το άρθρο 152 ούτε με το άρθρο 153 παράγραφος 5. Άρθρο 152 είναι μια γενική διάταξη που δεν αποκλεί την ανάγκη λήψης περαιτέρω ή μάλλον εξειδικευμένων μέτρων. Αλλά αυτή η διάταξη δεν δημιουργεί κάποια ουσιαστικά δικαιώματα για τις κοινωνικές πλευρές. Το άρθρο 153.5 αφορά το περιεχόμενο των μέτρων που μπορούν να υιοθετηθούν με βάση το άρθρο 153 στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Άρα αυτά τα, τις αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί λοιπόν με βάση το άρθρο 153. Οι κοινωνικέ πολιτικές φυσικά δεν θα πρέπει να παραβλέπονται, χρειάζεται να ληφθούν υπόψη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ως επιπτώσεις του άρθρου 153 του 5 μέτρα δεν, έχουν, δεν μπορούν να ληφθούν σε ό,τι αφορά τους ε, μισθούς τα μέτρα που το πήρε με βάση το 122 προβλέπουν τις προϋποθέσεις που συνδέονται με την χορήγηση βοήθειας. Και αυτό αναφέρεται ρητά στο 122.2. Δεν υπάρχει λοιπόν νομικό ζήτημα. Σε... Και επαναλαμβάνω ότι οι συνθήκες που αναφέρονται στο πρόγραμμα καλύπτουν ένα ευρύ τομέα πολιτικών, περισσότερες ε, εξ αυτών είναι οικονομικής φύσης και είναι θέσεις που συμφωνήθηκαν με το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος η Κομισιόν να γνωρίζει ότι οποιοδήποτε ε, πρόγραμμα ε, βοήθειας έχει οικονομικές ε, επιπτώσεις ε, αλλά οι διάφορες προϋποθέσεις έχουν ως στόχο να περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει η κρίση στην χώρα μέλος. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Για διαδικαστικό ζητάτε το λόγο. Διαδικαστικό και Ντερόσα. Μια διευκρίνηση διότι υπάρχει αντίφαση σε αυτά που είπε η Κομισιόν. Κοιτάξτε, έχει λήξει η συζήτηση κύριε Ντερόσα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να θεωρήσουν ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις ε, στην ε, απάντηση του Επιτρόπου. Μεστόση περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της Μεσητής Διατάξεως. Όχι, όχι, έχει ολοκληρωθεί, έχει κλείσει η συζήτηση κύριε Ντερόσα διαδικαστικό. Πείτε μου σε ποιο άρθρο του κανονισμού αναφέρεστε. Θα θέλω να σας ζητήσω το εξή. Όταν έχουμε έναν επίτροπο εδώ στο Κοινοβούλιο και αφενός δηλώνει ότι η Ιρλανδία δεν έρχεται καμία επιβολή για να μειώσει του μισθού και τα τροπή στο κοινωνικό, το κοινωνικό τη σύστημα και ε, ε, νομίζω όμως ότι αυτά είναι ε, αιρεσιμότητες ε, για να μπορέσει να διακόπτει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ, γνωρίζετε ότι σας συμπαθώ και είμαι ιδιαίτερα ευγενής μαζί σας, αλλά δεν μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε συζήτηση από την αρχή. Πρέπει να σεβαστούμε την ε, θέση σας όπως σεβόμαστε και τη θέση του Επιτρόπου έχει δικαίωμα στο να θεωρήσετε πως υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της μέσης διατάξεως που αφορά την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Είναι ερώτηση προφορική που προέρχεται από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, Ασφάλειας και Τροφή Και